Έχουμε μια σειρά από ε, ανακοινώσεις. Υπάρχουν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Υπάρχει κάποια παρατήρηση? Όχι. Εκ των προτέρων εγκρίνονται τα πρακτικά. Έχετε διαδικαστικό παρακαλώ. Σας ακούμε. Ήθελα να μιλήσω επί του προσωπικού γιατί εδώ ακούστηκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Η κυρία Τσίμερ προκειμένου να στηρίξει την πρόταση για να μπει στην, στην ατζέντα το θέμα της αύξησης του μεταναστευτικού μίσους και της βίας χρησιμοποίησε σαν αιτιολογία ότι στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αντιρατσιστική πορεία από το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Ή δεν το τι έγινε στην Αθήνα ή είπε ψέματα. Γιατί στην Αθήνα ήταν μια επέτειος τιμής και μνήμης για τρεις έλληνες ήρωες αξιωματικούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το 1996 και στα ήμια. Και αυτή την εκδήλωση φυσικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την απαγόρευσε. Σας ευχαριστώ. Καταγράφουμε αυτή την πληροφόρηση. Η διάταξη αναφέρει ότι θα έχουμε την κοινή συζήτηση